Ανατώθηκε η συζήτηση. Η επόμενη σύνοδος θα λάβει χώρα αύριο 5η 27 Φεβρουαρίου 2014 από τις 8.30 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Η μερίσια διάταξη δημοσιεύτηκε και είναι διαθέσιμη στην σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε διακόπτεται η συνεδρίαση. Καλώς σας βράδυ.